ανακοίνωσή της στα μέσα Οκτωβρίου θα επανέλθει για τα θέματα αυτά και θα μας βοηθήσει πολύ η έκθεση σας κύριε Γκέρεν σε αυτή την ανακοίνωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε και ευχαριστούμε και τον εισηγητή μας τον κύριο Γκέρεν. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση Φρανσίσκο Σόσα Βάγνερ για την ενεργειακή υποδομή και τις προτεραιότητες το 2020 και μετέπειτα. Κύριε Σόσα Βάγνερ, έχετε το λόγο. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πρώτα τους σκεώδεις εισηγητές για την καρποφόρα συνεργασία. Και το ίδιο το λέω και για τους υπόλοιπους συναδέλφους της Επιτροπής μου στο Κοινοβούλιο. Πριν από 60 χρόνια δημιουργήθηκε η ΕΚΑΧ δεν έχουμε καλύτερη ευκαιρία για την, να γιορτάσουμε αυτήν την επέτειο από το να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για την ενεργειακή υποδομή, τη μελλοντική ενεργειακή υποδομή της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει ορίσει με σαφήνεια την μελλοντική, ενεργειακή της υποδομή. Μιλάει για αυτάρκεια, εναλλακτικές ενέργειες, διαφοροποίηση της τροφοδότησης. Στην θήκη της Λισαβόνας έχουμε έναν τίτλο που, τον 21, το κεφάλαιο 21 που αφορά στην ενέργεια όπου αναφέρονται όλες οι δεσμεύσεις που ανέφερα όπως επίσης και το θέμα της, ο στόχος της διασύνδεσης των ενεργειακών υποδομών. Πρόκειται για δίκτυα τα οποία είναι κακώς διασυνδεδεμένα. Εμείς έχουμε μεγάλη αύξηση αιωλικής, παραγωγής αιωλικής ενέργειας στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακής ενέργειας στη Νότια Ευρώπη. Έχουμε άλλα κατεπήγοντα ζητήματα όπως το θέμα των σημείων φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πρέπει να δημιουργήσουμε νέα δίκτυα, νέες συνδέσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον να προχωρήσουμε στον ορισμό των απαραίτητων υποδομών. Πρώτον, ορίζοντας τα κριτήρια επιλογής σχεδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Β καταργώντας τα, τις, ενεργειακά, τις, ε, τις απομονωμένες παραγωγές ενέργειας. Θα πρέπει να χορηγήσουμε άδειες στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν δίκτυα. Δεύτερον, συνεργασία, ε, τέταρτο, συγγνώμη, συνεργασία για την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη δημόσια ενίσχυση, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, η οικονομία και τα ευφύ δίκτυα είναι το κεντρικό σημείο του νέου σχεδίου που εσωματώνουμε εδώ στην έκθεση. Διότι θεωρώ ότι με τη μείωση της ζήτησης ενέργειας θα μειώσουμε και την εξάρτηση από τις εισαγωγές και αυτό με όλες τις επιπτώσεις της ανάγκης υποδομής. Εμείς ε, στην έκθεση μιλήσαμε για το θέμα των αδειών για, ε, για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των έργων. Βέβαια, πολλά σχέδια ε, κολλάνε διότι ο πληθυσμός, ε, ο κόσμος δεν τα θέλει, δεν θέλει να βλέπει ε, πύργους, ή ε, ε, ε, ηλιακούς θερμοσυσσωρευτές. Πρέπει να τους πείσουμε και θα πρέπει μέσα σε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους να, να εμπλακούν όλοι. Χρειάζεται επίσης να έχουμε ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα χρηματοδοτείται σταθερά. Μέχρι τώρα η ενεργειακή πολιτική της Ένωσης τόσο εκτός και εντός της Ένωσης δεν είχε την ευρωπαϊκή πρόθεση. Η Ευρώπη θα πρέπει να μιλάει με μία και μόνη φωνή η οποία θα είναι ενιαία διότι από την ενεργειακή μας αδυναμία θα πρέπει εμείς να βγάλουμε δυνάμεις για να δημιουργήσουμε μια νέα Ευρώπη ενεργειακώς δυνατή η οποία σε αυτήν την επέτειο θα είναι και η, ε, η διάδοχος της ΕΚΑΧ που αποτελεί και την κούνια στην οποία γεννηθήκαμε. Βλέπω διάφορους που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Κάρινς ε, θα πάρει πρώτος τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι είμαστε όλοι ε, συνηθισμένοι να έχουμε την ελευθερία επιλογής. Όταν διαλέγουμε το σαπούνι μας, την τηλεόρασή μας, ε, ε, τον πάροχο υπηρεσιών για τηλεφωνική μας γραμμή, και ως ε, καταναλωτές <coughs> έχουμε το δικαίωμα να ε, επιλέξουμε τη χαμηλότερη τιμή ή την υψηλότερη ποιότητα, διότι ισχύουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Συχνά όμως ε, δεν υπάρχει επιλογή για την, παροχή, για την ηλεκτροδότηση και την παροχή φυσικού αερίου. Γιατί, διότι χωλένουμε στην διασυνδεσιμότητα των δικτύων για να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ενιαία αγορά για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Με αυτή την έκθεση διευκρινίζουμε πλέον ότι είναι δικαίωμα των πολιτών να έχουν επιλογή όχι μόνο όταν διαλέγουν σαπούνι και σαμπουάν αλλά και όταν αγοράζουν ενέργεια. και θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ναι, τη μέγιστη δυνατή επιλογή στη χαμηλότερη δυνατή ε, τιμή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο εξυγχρονισμός της ενεργειακής υποδομής ε, έχει ιδιαίτερη σημασία για να έχουμε βιώσιμη και ευφυή ανάπτυξη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη στρατηγική 2020 και να κατοχυρώσουμε την ενεργειακή ασφάλεια. Ε, πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη πρόκληση και μέσα στα κανονιστικά συστήματα υπάρχουν διατάξεις που πρέπει να βελτιωθούν κυρίως σε σχέση ε, με τα πλέον καινοτόμα προγράμματα ή τη διαχείριση του κινδύνου και προγράμματα κυρίως που αναφέρονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις εξόγους απόκεντρες περιφέρειες. Ε, θα πρέπει λοιπόν όλοι οι ενδιαφερομένοι να εμπλέκονται στην εκπόνηση του προγράμματος γιατί έτσι εξασφαλίζουμε τα βέλιστα δυνατά αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν μια ρεξικέλευση προσέγγιση και στον ενεργειακό τομέα, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές διαστάσεις του ζητήματος και θα πρέπει μέσω μακροπρόθεσμα να κατοχυρώσουμε τον ασφαλή ενεργειακό ανεφοδιασμό των πολιτών ε, με βιώσιμο τρόπο και σε προσιτές τιμές. Σας ευχαριστούμε. Κύριος Νικολάσικ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει τη νομική βάση για την ανάπτυξη της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σωστά για να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε και να βελτιώσουμε τη διασύνδεση, τις διασυνδέσεις και να βελτιώσουμε τις υποδομές των δικτύων ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να επιτύχουμε την πολιτική που έχουμε ορίσει ως στόχο για το 2020. Μέσω των πολιτικών συνοχής ε, μπορούμε επίσης να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία δίνει νέες δυνατότητες διαμεθοριακής συνεργασίας, ούτως ώστε να έχουμε διασύνδεση τοπικών και περιφερειακών πηγών ενέργειας και μεγάλων ενεργειακών δικτύων. Ο συντονισμός των υποδομών και των έργων ε, ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ε, αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων και για την επίτευξη ε, ε, της διασύνδεσης. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Φιγκερέιντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να τονίσω τη σημασία που έχει η ανάπτυξη της ενεργειακής παραγωγής και πόσο σημαντικό είναι να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές μέχρι το 2020 αν όχι και παραπάνω. Αλλά η ενέργεια είναι ένα στρατηγικό τομέα και απαιτούνται υψηλέ επενδύσει και άρα οι χώρε και οι περιφέρειες που έχουν οικονομικέ δυσκολίε δυσκολεύονται επίση να ακολουθήσουν τι αλλαγέ εξού και η ανάγκη ε, μέγιστου εξυγχρονισμού ναι μένα, αλλά προσοχή γιατί μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Να πληγούν τα ασθενέστερα στρώματα ακόμη περισσότερο χρειάζεται χρειάζονται δημόσιε ε, πολιτικέ υπεύθυνε ε, στον τομέα της ενεργειακή πολιτική, ε, ούτω ώστε συγγνώμη, να εξασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση ανεξαρτήτω όρων και προποθέσεων που ισχύουν για κάθε χώρα, για κάθε πολίτη. Δηλαδή χρειαζόμαστε πολιτικέ και υποδομέ που να καλύπτουν και τι περιοχέ που υστερούν. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση στην ενέργεια και θα παρεμποδίσουμε την διόγκωση της ενεργειακής ε, για να μην στερηθούν το ηλεκτρικό και τη ζέστη ε, εκατομμύρια νοικοκυριά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Κέλλη τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον εισηγητή για την ε, έκθεση αυτή διότι είναι απολύτω ε, καθοριστική σημασία για αυτό που θα κάνουμε μέχρι το 2020. Ε, πρέπει να υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Είναι καιρός. Ε, πρέπει να υπερασπιστούμε όχι τα παγκόσμια συμφέροντα, αλλά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ε, και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη συνολική η παγκόσμια ανάπτυξη. μέχρι το 2050 λοιπόν θα πρέπει να υιοθετήσουμε τα μέτρα για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια για την ενέργεια αιωλική ενέργεια, για την ε, βιοθερμική ενέργεια, όλες τις μορφές, τις, ε, ε, τις, όλες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ε, διότι τα ορεικτά καύσιμα, η εξάρτηση από τα ορεικτά καύσιμα θα πλήξουν την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε, να βρούμε την αλλακτική λύση για να την εξαγάγουμε στη συνέχεια στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει την αρχή της οικοδόμησης μιας μια ενεργειακή κοινότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέτρα που ανακοινώνεται τώρα θα εφαρμόζονται και στην περίοδο μετά το 2020. Δείτε τι προσπάθειες πρέπει να γίνουν για να αναβαθμιστούν οι ενεργειακές υποδομές ε, μέχρι το 2020 και μετά τα ενεργειακά δίκτυα του σήμερα δεν είναι ε, σε θέση από πλευράς τεχνολογίας ε, να διανύμουν νέες μορφές ενέργειας. Χρειαζόμαστε μια φρέσκια νέα προοπτική συνολικότερα στον ε, τομέα της ενέργειας και μέσα στην πολιτική που θα ακολουθήσουμε μέχρι το 2020 θα πρέπει να επικρατήσει ενάργεια και να δούμε ακριβώς πώς θέλουμε να σχεδιάσουμε τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Σα λοιπόν, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ακούσουμε τώρα την Επίτροπο ε, Μάλμστρομ για να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ αξιότιμοι βουλευτές, ε, εισηγητά. Ε, καλωσορίζουμε την ε, έκθεση πρωτοβουλίας για τις προτεραιότητες, για τις ενεργειακές υποδομές για την περίοδο 2020 και μετά. Φυσικά είναι η ύψιστη προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και τους κοιόδους εισηγητές για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Οι ενεργειακές υποδομέ είναι στην καρδιά του τομέα χωρίς σε τέτοιε υποδομέ, προηγούμενε τεχνολογίε δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε του ενεργειακού μα ε, στόχου. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να μεταρρυθμιστεί άρδιν το ενεργειακό μα σύστημα, το οποίο συνεπάγεται και μεγάλε προκλήσει, αλλά και μεγάλε νέε δυνατότητε για την παραγωγή και την κατανάλωση τη ενέργεια. Οποιοδήποτε μελλοντικό σενάριο προβλέπει ότι, μάλλον αποδίδει καταλητικό ρόλο στι ενεργειακέ υποδομέ για την υλοποίηση των στόχων. Στοκχόλμη. Λοιπόν, το Φεβρουάριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για λόγους αλληλεγγύης, για να είναι διαλειτουργικά τα συστήματα, για να έχουμε ε, εναλλακτικές ε, οδούς ανεφοδιασμού, ε, εναλλακτικές πρώτες ύλες. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτές τις αλλαγές για να μπορέσουμε να επανασχεδιάσουμε τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας των δικτύων και γι' αυτό είναι εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα. Έχουμε ήδη εγκρίνει την ανακοίνωσή μα ε, για τη μελλοντική ενεργειακή πολιτική. Θα ε, συνεχίσουμε ε, να επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους για να καλύψουμε τις εξής ανάγκες. Ε, τα δίκτυα υπερακτίως στη Βόρεια Θάλασσα συγκεκριμένα έχουμε μεγάλες δυνατότητες και μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης. Να διαφοροποιήσουμε τις οδούς παροχής φυσικού αερίου οικοδομώντας τον νότιο διάδρομο. Διασύνδεση στην νοτιοανατολική Ευρώπη ούτως ώστε να δημιουργήσουμε νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ρέει αυτονότερο το φυσικό αέριο στην περιοχή αυτή. Επίσης, ε, η ε, αγορά πετρελαίου και φυσικού αέριου δεν πρέπει να περιορίζεται τις ενεργειακές νησίδες. Ε, θα πρέπει να είναι απόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως σε προβληματικές περιοχές όπως είναι η Ανατολική Ευρώπη. Θα πρέπει τώρα να περάσουμε στη δράση από τα προγράμματα, από τα προσχέδια, να περάσουμε στη διαβούλευση, στην αδειοδότηση, στη χρηματοδότηση και την επιτόπου οικοδόμηση. Και γι' αυτό η επερχόμενη νομοθετική μας πρόταση για τις ενεργειακές υποδομές θα έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ένα βασικό στοιχείο για την εφαρμογή των στόχων περί ενεργειακών υποδομών είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Εκτιμάται ότι άνω των 200 δις ε, χρειαζόμαστε τα επόμενα χρόνια. Ε, ε, και δεν πρόκειται να ε, προκύψουν από μόνες τους οι επενδύσεις. Πέρσι εγκρίθηκε, συγγνώμη, χτες εγκρίθηκε η πρότασή μας για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014 2014-2029,1 9,1 δις θα διατεθούν για αυτό το σκοπό και έτσι αναγνωρίζεται η ανάγκη και ειδική χρηματοδότηση για τις ενεργειακές υποδομές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς μας στόχους ε, και να συνεχίσουμε ασφαλή αναφοδιασμό με ανταγωνιστικό τρόπο για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, καλωσορίζουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, όπως φαίνεται μέσα στο ψήφισμά σας, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, ε, αναγνωρίζουμε τις συστάσεις που συμπεριλαμβάνει η έκθεση και τις επικροτούμε, κυρίως ως προς την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τα προγράμματα ενεργειακών υποδομών, την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και καλύτερη εμπλοκή των άμεσα ενδιαφερόμενων και επίση η προώθηση διασυνοριακών υποδομών και χρηματοδότηση. Ε, θα τα λάβουμε όλα αυτά δεόντως υπόψη για να εκπονήσουμε την τέταρτη νομοθετική πρόταση για την ανάπτυξη, τη μελλοντική ανάπτυξη των ενεργειακών ε, υποδομών. Μπορείτε να αναμένετε την ανακοίνωσή μας στο φθινόπωρο. Σας ευχαριστούμε για την πρόταση και σας ευχαριστούμε κυρίως ε, για την υποστήριξή σας, τόσο ώστε να έχουμε τα, ενεργεια... τα ενεργειακά δίκτυα που χρειαζόμαστε για το 2020 και μετά. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε και ευχαριστώ και τον εισηγητή τον κύριο Σώσα Βάγκνερ και τώρα... Περνούμε στην επόμενη έκθεση που είναι η έκθεση του κυρίου Ντερόσα, κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Παρακαλώ.